So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Δεν είμαστε πολλοί. Αλλά όλο και κάποιος φαντάζομαι θα έρθει. Είναι σημαντική η συζήτηση που έχουμε μπροστά μας. Και καλώς ορίζω τον κύριο Ντανιέλε Βιώτη, τον ε, εισηγητή του προϋπολογισμού για το 2019. Ξέρω κύριε Βιώτη ότι έχετε να επισκεφτείτε όλες τις επιτροπές. Έχετε αρκετά σκληρή δουλειά μπροστά σας. Και ελπίζω να μας παρουσιάσετε σήμερα τις προτεραιότητες σας για το 2019. Και θα ακούσετε τις δικές μας προτεραιότητες ε, από την οπτική γωνία του πολιτισμού της παιδείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος ε, Μαΐου θα παρουσιάσει το σχέδιο προπολογισμού και το Μάιο θα δημοσιευθούν επίσης και οι προτάσεις για το πρόγραμμα των ε, υπολείπων οργάνων για το 2019, αλλά θα αφορούν και την περίοδο μετά το 2020. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά στον εισηγητή κύριο Λόκιγκαρντ, ο οποίος ασχολείται με θέματα προϋπολογισμού. Μετά θα λάβουν το λόγο τα υπόλοιπα μέλη και σχεώδες συζητητές, όμως ε, κύριε Ντάνιελ Λεβιώτη έχετε το λόγο για περίπου πέντε λεπτά. Και χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε να σας πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, και φυσικά σας ευχαριστώ και για την ε, φιλοξενία. Ε, ουσιαστικά κάνω ένα γύρο και επισκέπτομαι τις διάφορες επιτροπές και μαθαίνω πάρα πολλά. Μαθαίνω και τους διάφορους τρόπους εργασίας και τις δραστηριότητες των επιτροπών. Θέλω να πω δύο γενικά πράγματα για τον προπολογισμό, περισσότερο μεθοδολογικά παρά θέματα ουσίας. Στη συνέχεια θα μπω στα θέματα ουσίας πολύ σύντομα, γιατί φυσικά συμφωνώ απόλυτα με πολλές από τις σκέψεις που έχουν εκφραστεί και από Ιταλούς ε, συναδέλφους σε σχέση με το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, βάσει των οποίων ε, θα κινηθεί και η σημερινή συζήτηση. Για την μέθοδο, όπως σας είπα, εσείς ε, γνωρίζετε πόσο σφιχτός είναι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είναι πολύ πολύπλοκο να κινηθούμε και το λέω και για την Επιτροπή Πολιτισμού. Είναι λοιπόν δύσκολο να κινηθούμε με φαντασία και να εκφράσουμε ε, ουσιαστικά το στοιχείο της φαντασίας που μπορεί να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα προπολογισμό. Αυτό συνδέεται και με ένα άλλο στοιχείο στο οποίο θα επιστρέψω στη συνέχεια. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο συνεχίζει να ζητά νέα προγράμματα από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητά λοιπόν να υλοποιηθούν νέα προγράμματα χωρίς να θέλει να χρηματοδοτήσει αυτές τις νέες πολιτικές και αυτά τα νέα προγράμματα. Έτσι λοιπόν είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση γιατί όπως ε, ξέρετε δεν πολλαπλασιάζονται τα χρήματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ούτε ο, η Επιτροπή Προπολογισμού, το εισηγητή σας, ε, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει ε, να ε, εγκαταλείψει προγράμματα τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν σημειώσει επιτυχία και στα οποία εμπιστεύονται οι πολίτες και τα διάφορα όργανα για τα επόμενα έτη. Έκανα αυτή την ε, εισαγωγή που ήταν πιο μακροσκελής από ό,τι ήθελα, αλλά το έκανα για να πλαισιώσω το γενικό ζήτημα του προπολογισμού. Ακόμη και θα δούμε και στη συνέχεια το τελευταίο θέμα της ε, συνδιαλλαγής. Όπως και η προκατοχή μου, θα συνεχίσω να εργάζομαι προκειμένου να υπάρξει όσο δυνατόν μεγαλύτερη συνένεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προπολογισμό, γιατί πιστεύω ένα πολύ ισχυρό και ενωμένο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια ευρεία πλειοψηφία θα είναι πιο ισχυρό την στιγμή της συνδιαλλαγής με το Συμβούλιο. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια διευρυμένη συνένεση όχι μόνο για τις ε, πολιτικές ομάδες, ε, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ομάδες, αλλά και σε ό,τι αφορά τις διάφορες επιτροπές. Έτσι λοιπόν, ε, τα αντιζεντεράτα των διάφορων επιτροπών θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω στο δυνατόν περισσότερο. Φυσικά θα ακούσω ποιες, ποια είναι τα κυριότερα αιτήματα και θα υλοποιήσω τις προτάσει. Σα Υπάρχει φυσικά ένα ζήτημα που αφορά το Erasmus Plus, το Erasmus In. Από πολιτική και συμβολική σκοπιά είναι το πιο, το πιο σημαντικό στοιχείο. Στις κατευθυντήριε γραμμές που παρουσίασα και ψηφίσαμε το Μάρτιο στην Ολομέλεια, θα είδατε ότι εκεί είχα γράψει ότι σκόπευα να ζητήσω το διπλασιασμό του προϋπολογισμού της χρηματοδότησης για το Erasmus+. Τώρα για τη δημιουργική Ευρώπη. Συμφωνώ ότι υπήρχαν ε, προβλήματα υποχρηματοδότησης. Ε, περίπου χάθηκε το 20% και από την ε, Δημιουργική Ευρώπη και από το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Κατόπιν το πρόγραμμα της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών. Συζήτησα για αυτό το πρόγραμμα και με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Δημιουργήθηκε μία νέα γραμμή, αλλά δεν έχουν καταναμηθεί πόροι για αυτή τη νέα γραμμή προπολογισμού. Κοιτάξτε, είναι κάτι άχρηστο. Δεν θέλω να πω το κορίδι του πολίτε, αλλά είναι κάτι άχρηστο. Κατόπιν τώρα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Φυσικά το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν θα πω σε λεπτομέρειε. Αλλά, όπω είπα στην αρχή, θα αναφερθώ εκ νέου σε αυτό το σημείο. Ε, στα νέα προγράμματα θα πρέπει να αντιστοιχούν νέοι πόροι. Και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να σκεφτούμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, που είναι ε, ένα project όλης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, θα είναι ένα πρόγραμμα το, από το οποίο θα ε, λειτουργήσει με την αφαίρεση πόρων από υφιστάμενα προγράμματα. Αυτές είναι λοιπόν οι κατευθυντήριες γραμμές βάσει των οποίων θα κινηθούμε. Φυσικά υπάρχουν ε, και άλλα θέματα, όπως ε, παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού δεν είναι επαρκής η ούτε εκεί και προσπαθήσαμε να έχουμε ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού, αλλά δεν ε, τα καταφέραμε λόγω ε, του ότι είναι σφιχτός ο προπολογισμό, όπως σας είπα. Και βέβαια θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να έχω την υποστήριξη της δικής σας επιτροπής, όχι μόνο σήμερα, με τη δική σας γνωμοδότηση, αλλά και τους επόμενους μήνες, όταν θα βρισκόμαστε σε κρίσιμη χρονική συγκυρία. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως η στήριξη της Επιτροπής μας για όλα τα θέματα τα οποία στην αρμοδιότητα μας είναι δεδομένη. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε σύντομα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και δεν μπορώ να πω ότι μας εξέπληξα. Ίσως μας ενόχλησε λίγο η στάση του Συμβουλίου, των κρατών μελών δηλαδή, που δεν είναι έτοιμα να διαθέσουν νέους πόρους για αυτή την πρωτοβουλία. Και στην περίπτωση αυτή ε, τα, οι νέοι πόροι δεν σημαίνουν κονδύλια που μεταφέρονται, δεν σημαίνουν κονδύλια που θα επιβαρύνουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να συσταθεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Βέβαια, είναι ε, αυτονόητο ότι τα νέα μέτρα θέλουν και αντίστοιχους νέους πόρους. Είναι λοιπόν ε, δυσάρεστο ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να διαθέσουν κονδύλια. Το πρόγραμμα Erasmus SIN ε, είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές μας, το αναφέρατε κι εσείς. Στην Γενική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ζητούμε τριπλασιασμό των πόρων στην Επιτροπή μάλιστα έχει γίνει λόγος για πολλαπλασιασμό των πόρων και κάποια κράτη-μέλη ζήτησαν δέκαπλασιασμό. Και μάλιστα ακούσαμε πολλές έτσι υποσχέσεις διανθισμένες με όμορφα λόγια, αλλά ο διπλασιασμός που μας υποσχέθηκαν δεν είναι, ο πρόεδρος της Επιτροπής δεν είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα ιδιαίτερα όχι μόνο σε ό,τι αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη. Το 2019 και το 2020 θα χρειαστεί χρηματοδότηση ε, από το Πουδουπού και πιστεύω ότι θα είναι έτσι, πολύ δύσκολε οι συζητήσει που θα ακολουθήσουν. Σα ευχαριστούμε όμω πάρα πολύ που ήρθατε, μα παρουσιάσατε την κατάσταση στην Επιτροπή Πολιτισμού θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Μόρτεν Λόκεγκαρτ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι συμφωνώ και εγώ με τα περισσότερα που όσα είπατε. Η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής μου δίνει ιδιαίτερη εμπειρία συνήθως υπάρχει μεγάλη συνένεση για αυτά τα θέματα και ως ε, παλαιότερο μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού να πω ότι αισθάνομαι πως αντιγράφουμε απόλυτα αυτά που γίνονται εκεί. Και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση εδώ. Άκουσα αυτά που είπατε κύριε Βιώτη και θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη στήριξη που μας ε, δείχνετε εσείς, διότι αναφέρατε τις ίδιες προτεραιότητες που έχουμε και εμείς. Και χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε στα ίδια μήκη κύματος. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ καλή αρχή αυτή. Ο προπολογισμό του 2019 είναι κατά κάποιον τρόπο πρόδρομος του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και δεδομένου ότι δεν έχουμε δει ακόμα κάποιο σχέδιο προϋπολογισμού, αλλά ένα προσχέδιο, παρατηρώ ότι υπάρχουν κάποια γενικά σχόλια για την ε, οριοθέτηση προτεραιοτήτων και μετά κάποιες έτσι γενικές αναφορές ε, στις ευρύτερε προτεραιότητες. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με ορισμένα προγράμματα και ορισμένα έργα τα οποία έχουν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό προέκυψε στις τελευταίες συζητήσεις και να σας πω ότι δεν γνώριζα ότι υπάρχουν τόσα πολλά διαθέσιμα δισεκατομμύρια ευρώ για άλλα προγράμματα όμως. Μου φάνηκε έτσι αρκετά περίεργο και θα ήθελα λοιπόν να αναφερθούμε λίγο στο θέμα αυτό της διαχείρισης των ε, τόσων δισεκατομμυρίων ευρώ. Νομίζω πως πρέπει να δώσουμε προσοχή σε αυτό. Θα επανέλθω όμως. Στην ουσία, χρειάζεται μια γενικότερη εικόνα στο πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για τον πολιτισμό. Και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το σημείο 1, όπου αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση του Εράσμους ΣΥΝ, Όπως είπατε και εσείς, οι γενικές γραμμές τονίζουμε επίσης στο σημείο 2 την αξία της δημιουργικής Ευρώπης, του Creative Europe, μετά την ανάγκη να εξασφαλιστούν κονδύλια για το Euronet. Ίσως θα μπορούσατε κι εσείς να το λάβετε υπόψη, γιατί είναι κάτι που έχει συζητηθεί αρκετά στην Επιτροπή. Το Euronet είναι ένα πρόγραμμα το οποίο από άποψη χρηματοδότησης είχε αρκετά προβλήματα. Μάλιστα αμφισβητήθηκε και η ίδια η βιωσιμότητά του εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπω όμως τώρα ότι ξεκαθαρίζει λίγο το τοπίο, είναι θετικές οι εξελίξεις. Θα ήθελα λοιπόν να δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στον ερχόμενο προϋπολογισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να επιβιώσει αυτό το πρόγραμμα και μάλιστα φροντίζει να παρέχονται και οι πόροι γι' αυτό. Διαφορετικά, γιατί να το έχουμε ανοιχτό, ας το κλείσουμε. Και μάλιστα να σας πω ότι πολλοί αποχωρούν αυτό το πρόγραμμα, το εγκαταλείπουν ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν πόροι. Χρειάζεται λοιπόν να βρεθούν αμέσως χρήματα. Μετά, στο σημείο 4 τονίζουμε την αξία των πολιτών της Ευρώπης και στο σημείο 5, όπως είπα και πριν, ζητάμε από την Επιτροπή να βελτιώσει τις συνέργειες ανάμεσα στα προγράμματα με θέμα πολιτισμό και εκπαίδευση. Ίσως δείτε ότι αναφέρεται το ποσό των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ από 11 σε 13. Από 7 σε 13. Χρειάζεται να δούμε πιο οργανωμένα το θέμα της χρηματοδότησης από μια γενικότερη οπτική γωνία. Κάτι ακόμα πριν σταματήσω να πω πως λάβαμε κάποιες πληροφορίες από την Επιτροπή για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, Europe for Citizens. Όπως γνωρίζετε, θα μειωθεί ο μειώθηκε ο προϋπολογισμός κατά 750.000 ευρώ για να χρηματοδοτηθεί μια ε, άλλη πρωτοβουλία, το Citizens Initiative το, στην τελευταία επικαιροποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος αναφέρεται ότι θα μειωθεί ο προϋπολογισμός κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο 2019 μέχρι το 2020 για αυτήν την πρωτοβουλία πολιτών. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Πρώτον, μειώνεται ο προϋπολογισμός του Ευρώπη για τους πολίτες κατά 5%. Είναι ουσιαστική μείωση για ένα πρόγραμμα που ήδη υποχρηματοδοτείται, όπως είπατε κι εσείς. Ήδη αυτό το θέμα έχει αναφερθεί για τον προπολογισμό του 2018. Έπειτα, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις ε, δεν αιτιολογούνται στην πρόταση της ε, Κομισιόν. Και ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θεωρεί ότι μετακινούνται με σωστό και νόμιμο τρόπο κονδύλια, έτσι, όμως είναι θέμα αρχής πιστεύω. Δηλαδή, πώς εγκρίνονται πολιτικές αποφάσεις. Και εδώ υπάρχει θέμα αρμοδιότητας Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να σας επιστήσω την προσοχή σε αυτά και θα σταματήσω εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μόρτεν. ισχυώδη ηγητές τώρα. και τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ξεκινώντα να πω ότι με μεγάλη χαρά άκουσα τόσο είχατε να πείτε για το Erasmus Plus. Ανεξαρτήτως του ότι δεν τριπλασιάστηκαν αλλά διπλασιάστηκαν τα ποσά, εμείς ελπίζουμε να τριπλασιαστούν, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από τα λόγια σας. Πριν από χρόνια είχαμε αγώνα να προστατεύσουμε το ίδιο το πρόγραμμα που μόνο θετικό αντίκτυπο έχει. και που, δεν δεν, να έχει ολοκληρώσει το έργο του, όπως ορισμένοι έλεγαν. Τώρα ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να ενισχυθεί. Ο διπλασιασμός λοιπόν των κονδυλίων για το Erasmus Plus νομίζω μπορεί να μας ικανοποιεί όλους. Επίσης μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την ιδέα το Δημιουργική Ευρώπη να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και να πάρει το δικό του δρόμο. Ήταν χρήσιμη σαν ιδέα, πρέπει να ενισχυθεί τώρα. Στο Ευρώπη για τους πολίτες. Θα ήθελα να σταθώ, αλλά πρώτα θα πω δύο λόγια για το προγράμματα μαζί. Για να εξασφαλίσουμε ένα 11 και 16% μόνο στη χρηματοδότηση, 90% των νέων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων θα στερηθούν τη δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα. Όταν ένα πρόγραμμα απορρίπτει όμως 30 έως 40% των αιτήσεων, γεννά αρνητικές εντυπώσεις. Γιατί θα είναι πολύ οι δυσαρεστημένοι από το πρόγραμμα. Πολλές αιτήσει που θα είναι και σωστές, θα πληρούν και τα κριτήρια και τους στόχους του προγράμματος, σε μεγάλο βαθμό μέχρι και 90% μπορεί να απορρίπτονται. είναι σαν να προσπαθούμε σε όρους πολιτισμού να χτίσουμε ένα αυτοκινητόδρομο που πρέπει να έχει μήκος χίλια χιλιόμετρα και να χτίσουμε μόνο τα 15. Το ίδιο και στον πολιτισμό λοιπόν. Ένα τέτοιο ποσοστό απόρριψη των ε, αιτήσεων. Το βλέπουμε ήδη. Ακόμη και αν τα ποσά δεν είναι τόσο σημαντικά στο σύνολο του προϋπολογισμού. Μιλούμε για κλάσματα του προϋπολογισμού και μάλιστα μικρά κλάσματα. Τα προγράμματα λοιπόν Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη για τους πολίτες δεν έχουν τη χρηματοδότηση που αξίζουν. Και δεν βλέπω να υπάρχει επαρκή συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ. Νίκοφ που αντικαθιστά τον κύριο Μουράνο. Ευχαριστώ, Πέτρο. Θέλω να συγχαρώ τους εισηγητές τις εκθέσεις και βέβαια εκπροσωπώ τον Λουίτζι Μωράνο, ο οποίος επισημαίνει ότι ήταν καλές οι γνωμοδοτήσεις, καλή βάση εργασίας, συμφωνεί με τον εισηγητή, με τους εισηγητές και επισημαίνει, ήδη το γνωρίζετε για ορισμένα θέματα, ότι πρέπει να Υπενθυμίσουμε την ανάγκη να ενισχυθεί το Erasmus Plus στην ε, αναθεώρηση του πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, η Δημιουργική Ευρώπη, η Ευρώπη των ε, πολιτών, υπενθυμίζει ο κ. Μωράνο, υποχρηματοδοτούνται και πρέπει τα δημοσιονομικά όρια να ε, ενισχυθούν για να χρηματοδοτούνται περισσότερα έργα. Είναι πολύ χαμηλή η απορρόφηση σε ορισμένα επίπεδα για το έτσι και τα ταμεία λέει ότι θα πρέπει να ενισχυθούν μέσα από αυτά ο πολιτισμός, η ο κλάδος της δημιουργίας, η προαγωγή της πολυγλωσσίας και των ποιοτικών θέσεων εργασίας και της αηφόρου ανάπτυξης. Αυτό δεν αναφέρεται. Ο κύριος Μόρκαν όμως γνωρίζει ότι είναι περιορισμένος και περιορισμένη και η, έκταση της γνωμοδότησης αναγκαστικά. Και θα καταθέσει τροπολογίες. Βεβαίως περιμένουμε την αξιολόγηση από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής των πιλωτικών έργων και των προπαρασκευαστικών δράσεων για να συζητήσουμε τα θέματα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για πολιτικές προτεραιότητες. Επίσης, ο συνάδελφο αναφέρεται σε ζητήματα αποφάσεων που ελήφθησαν πέρσι και φέτος και που θα έχουν αντίκτυπο στο προσεχές που δουπού και τι δεν συνδέονται καταρχήν με αυτό. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Αυτά έχει να πει ο κ. Μουρκάνο για το θέμα. Και ελπίζω να συνεργαστούμε όλοι μαζί με το πράγμα συνένεσης που απαιτείται. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Νεριάντα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον ε, εισηγητή και τον κύριο Βιώτη. Με χαρά σας βλέπω εδώ στην Επιτροπή του Πολιτισμού εκτός από την Επιτροπή Προϋπολογισμών στην οποία επίσης είμαι συντονίστρια. Πρέπει βεβαίω να αντιληφθούμε τι συνέπειε θα έχει και για, το, και για, την, ε, για τον πολιτισμό ο προπολογισμό του 19 αλλά και το Πουδουπού που επίση θα πρέπει να μα απασχολήσει. Εν γέννη είναι ευπρόσδεκτη η έκθεση, όντα μέλο και τη Επιτροπή των Προπολογισμών, παρακολουθώντα και τη δουλειά των άλλων επιτροπών. Ξέρω ότι ο καθένα έχει τι δικέ του προτεραιότητε. Δεν πρόκειται για την ε, μία κρίση, για την άλλη. Όλο και συμπιέστε προ τα κάτω η θέση τη δουλειά τη Επιτροπή Πολιτισμού. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τεράστια προσθέμενη αξία που έχουμε να προσφέρουμε με τον πολιτισμό και με την οικονομική ανταπόδοση που μπορεί να φέρει με το κέρδος το οικονομικό, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με την παραγωγή πολιτιστικού έργου. Υπάρχει αντίκρισμα οικονομικό που πρέπει να τονίσουμε. Είναι μια σοβαρή επένδυση, δηλαδή, επένδυση στον πολιτισμού και αυτό πρέπει να τονίσουμε. Και επίσης, σε δώσω δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει νομίζω κυρίως να μιλήσουμε για ισοδεμή πρόσβαση στον πολιτισμό, την εκπαίδευση για κάθε έναν, κυρίως αυτούς που για διάφορους λόγους κοινωνικούς ή άλλους βρίσκονται σε βιονεκτική θέση. Πρέπει να εισαχθεί και η διερμηνία στην γλώσσα των κοφών, στην οματική γλώσσα και στην ολομελία μας. Όσο δεν το έχουμε κάνει αυτό δίνουμε λάθος μήνυμα στους πολίτες εάν αυτό το εγκρίνουμε και δεν το υλοποιούμε όπως έχει συμβεί. Είναι πολύ μπερδεμένο το μήνυμα που αποστέλουμε. Αυτό λοιπόν έχω να πω για την Επιτροπή. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα πολλά. Αλλά μπορούμε να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στις δαπάνες και να εντοπίσουμε το πραγματικό οικονομικό αντίκρισμα των επενδύσεων μας, που είναι πολύ πιο σημαντικές ε, στους τομείς της Επιτροπής Πολιτισμού από ό,τι σε άλλες επιτροπές, γιατί χάρη στην ε, δημιουργία, χάρη στον πολιτισμό μπορούμε να βοηθήσουμε πολλούς να ξεφύγουν και από τη φτώχεια. Κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν πολλές άλλες επιτροπές με τη δουλειά Του Αυτό ελπίζω να το αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ τον εισηγητή, ευχαριστώ τον κύριο Βιώτη και πρέπει να πω ότι δεν καθόλου τη δουλειά που τον περιμένει. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τρούπελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα ήθελα συντομία να αναφέρω αυτό που είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Η πλειοψηφία αυτή της Επιτροπής πιστεύω ότι θέλει μεγαλύτερο προπολογισμό για το Erasmus Plus ε, και τη δημιουργική Ευρώπη. Ε, τώρα έχουμε ακόμα στον τριμερή διάλογο ε, το φάκελο για την υπηρεσία ελληνικής αυτά γιατί όλα τα προγράμματα μας αφορούν τα άτομα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, κοινωνική συμμετοχή και ε, καταλαβαίνουν οι πολίτες ε, τι κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Έχουμε λοιπόν πολύ ισχυρά επιχειρήματα υπέρ μας. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να πείσουμε τους υπουργούς οικονομικών αλλά και άλλους που ασχολούνται με τη γεωργία και τα ταμεία συνοχής. Όμως έχουμε πάρα πολύ καλά επιχειρήματα γιατί ξέρουμε τις Κυριακές όλοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα δικά μας επιχειρήματα για τη σημασία του πολιτισμού και την συμμετοχή των ανθρώπων και την ένταξή τους, ακόμη και των μεταναστών, μέσω του πολιτισμού. Στο επόμενο πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο, λοιπόν, θα είναι μεγάλη πρόκληση. Δεν έχουμε αρκετούς πόρους. Στο σημερινό δημοσιονομικό πλαίσιο και αν θέλουμε να ενδυναμώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, τότε ε, χρειαζόμαστε και αυξημένο προπολογισμό ε, από τους ίδιους πόρους ε, και χωρίς εκτόσεις. Και ξέρουμε ότι υπάρχουν φήμες στην Κομισιόν ότι ίσως τα προγράμματα μας δεν θα προβληθούν τόσο όσο θα έπρεπε. Πρέπει λοιπόν να, στείλουμε ένα σαφέ μήνυμα όταν θα συζητούμε τον επόμενο προπολογισμό ότι ο πολιτισμό είναι τόσο σημαντικός που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ε, να καλυφθεί μέσω των αρμοδιοτήτων άλλων επιτροπών και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε μεγάλη μάχη με το Συμβουλίο και την Κομισιόν. Σα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το συζητήσαμε και στη συνεδρία των συντονιστών και κατέστη σαφές ότι θα πολεμήσουμε με νύχια και με δόντια. έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτήν την ανάμειξη του πολιτισμού με άλλα προγράμματα. Ο κύριος Οφλίν έχει τώρα το λόγο. Να είστε σύντομος. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχα κάποιες ερωτήσεις στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρόεδρου Μακρόν την περασμένη εβδομάδα όπου από τη μία υποσχέθηκε περισσότερα χρήματα από τη Γαλλία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Βιώτη εάν έχετε περισσότερες λεπτομέρειες, αν έχουν αναλάβει τέτοιες ε, υποχρεώσεις και άλλα κρατημέλη και τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στους υφιστάμενους πόρους. Επίσης, ε, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μακρόν προσπάθησε να δώσει ένα στίγμα για να δημιουργηθεί αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και αρκετά από τα προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής σχετίζονται με αυτό. Υπάρχει γενικότερη επιθυμία να δημιουργηθεί αλληλεγγύη, σύνδεση μεταξύ των κρατών μελών. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα ανέβουν στην ε, στο κατάλογο των προτεραιοτήτων αυτά τα προγράμματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να κάνω μια παρατήρηση, επιτρέψτε μου, διότι νομίζω πως έχουμε ανακατέψει λίγο τις ε, συζητήσεις, έχουμε μπερδέψει. Οι δύο ημερήσεις διατάξεις που... Τα δύο σημεία της ημερήσιας διάταξης μάλλον που είχαμε σήμερα έτσι κάπως συγχέονται. Την τελευταία, την περασμένη εβδομάδα το Άρτε είχε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, Άρτε Europe Εκεί, να σας πω επί τη ευκαιρία του το Άρτε, είναι ένα κανάλι το οποίο δίνει έμφαση στον πολιτισμό. Αναφέρθηκε λοιπόν στο πρόγραμμα αυτό ένα πιλωτικό πρόγραμμα και μία προπαρασκευαστική δράση που έλαβε χρηματοδότηση τα προηγούμενα χρόνια και σκοπεύει να διαθέτει το πρόγραμμα του Άρτε σε έξι γλώσσες και όχι μόνο σε γαλλικά και γερμανικά όπως μέχρι τώρα, σε πολωνικά, ισπανικά, ιταλικά και αγγλικά πέρα από τις δύο γλώσσες που αναφέραμε. Το πρόγραμμα αυτό θα τελειώσει φέτος και θεωρώ πως είναι ένα εξαιρετικό έργο, μια πολύ καλή προσπάθεια. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε πώς αυτές οι προπαρασκευαστικές δράσεις θα λάβουν τη μορφή ε, προγραμμάτων τα οποία θα αγκυροβοληθούν στον προπολογισμό, θα τρέχουν συνέχεια. Γνωρίζουμε βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα προγράμματα που χρειάζονται χρηματοδότηση. Υπάρχουν, υπάρχει όμως η δυνατότητα ή θα έπρεπε έστω να υπάρχει, να δοθεί χρηματοδότηση και σε άλλα τέτοια πιλωτικά προγράμματα, όπως αυτό με το ARTE. Και ίσως στη γνωμοδότηση θα μπορούσατε να αναφέρετε ότι είναι επιθυμία μας να συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα πέρα από τις προπαρασκευαστικές δράσεις, να συμπεριληφθούν και μόνοι στον προϋπολογισμό. Να δούμε λοιπόν πώς θα καταφέρουμε Αυτά τα καλά, αποδεδειγμένα καλά προγράμματα πολιτισμικών ανταλλαγών στην Ευρώπη που μπορούν να φτάσουν μέχρι και στο 70% των Ευρωπαίων πολιτών θα σταθούν στα πόδια τους, θα λαμβάνουν την ε, κατάλληλη χρηματοδότηση. Είναι πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό και την ε, περασμένη εβδομάδα που επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις του Άρτε αυτό κατέστη σαφές. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον το επιθυμεί στον κύριο Βιώτη και θα κλείσουμε με τον κύριο Λόκιγκαρντ. Θα θέλατε το λόγο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, προσπαθήστε μέσα σε δύο-τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρίες ε, και κύριοι, κύριε Σιγητά, η Κομισιόν θέλει να σας ευχαριστήσει για την πολύ υποστήριξη ε, στα προγράμματα πολιτισμού νεολαίας ε, και παιδείας ε, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε στην ατόνα περισσότερα ωφέλη για τους δικαιούχους τους νέους, τους εκπαιδευτικούς κτλ. Ε, υπάρχουν έντονε διαπραγματεύσει, ε, όπω είπατε, και στα πλαίσια τη προετοιμασία του επόμενου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και τη προετοιμασία τη επόμενη νομική βάση. Εμεί ε, συμπιώνουμε του διάφορου πολυπλησιαστικού συντελεστέ που μπορούσαμε να ακούσουμε για διάφορα προγράμματα και κυρίω για το Erasmus Plus. Αυτά θα είναι πολύ σημαντικά για την προετοιμασία του προπολογισμού του 2019. Τώρα είμαστε στο δεύτερο ήμιση των προγραμμάτων από τι αρχέ του 2018 συνεχίζουν ε, τα προγράμματα να αναπτύσσονται σε πλήρη ταχύτητα και να παρουσιάζουν αποτελέσματα ε, με ένα ποσοστό εκτέλεση του προπολογισμού για τι επιχειρησιακέ επιστώσει κοντά στο 100%. Το ίδιο είχαμε και στο 2017 ω προ τη διαδικασία. Δυστυχώ δεν μπορώ να σα παρουσιάσω αριθμητικά στοιχεία για τον προπολογισμό, γιατί το Σώμα των Επιτρόπων δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση και δεν έχουν ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή ημερομηνίε για την απόφαση αυτή. Όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίε θα επανέλθουμε. Διαπιστώνουμε ωστόσο ότι στο επίπεδο του Erasmus Plus υπάρχει αύξηση των αναγκών ε, για τις πιστώσεις πληρωμών ε, επειδή στα κράτη-μέλη ε, οι εθνικοί οργανισμοί απορροφούν γρηγορότερα τις πιστώσεις από τα προηγούμενα έτη. Υπάρχει αυτή η διαπίστωση. Η επιτυχία των προγραμμάτων μα παρουσιάστηκε κυρίως ε, με τον εορτασμό ε, των 30 ετών ε, του Εράσμους. Βέβαια, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ζήτηση που δεν ικανοποιείται. Υπάρχει ε, λοιπόν ε, μια ε, μεγάλη ζήτηση όπως αναφέρονται και ίσως με περισσότερα κονδύλια θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε με περισσότερη ζήτηση, να υποστηρίξουμε περισσότερα project και να έχουμε περισσότερη κινητικότητα. Επίσης, ε, ε, σας ε, ευχαριστούμε για τα επιτεύγματα για τον περιπολογισμό του 2018 στο τμήμα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και κυρίως της κινητικότητας και της στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Επίσης είχαμε πρόσθετο προϋπολογισμό για την δημιουργική Ευρώπη. Ε, τα 2,5 εκατομμύρια θα τροφοδοτήσουν ε, τα σχέδια συνεργασίας δίνοντας έμφαση στην ένταξη των προσφύγων όπως είχατε ζητήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό δημοσιονομικό πλαίσιο, στο πλαίσιο των ε, διαπραγματεύσεων για τα μελλοντικά προγράμματα, η Κομισιόν ε, χαίρεται για τη μόνιμη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχουν επαρκή κονδύλια αυτά τα προγράμματα στους διάφορους τομείς δραστηριότητας. Επίσης, ε, χτες, ε, στην ομάδα παρακολούθηση στην Επιτροπή Προπολογισμού παρουσιάσαμε το Erasmus Plus και εκεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμού επέμεινε για να έχουμε ενδεχομένως ε, ε, επιτρία τριπλασιασμό του προϋπολογισμού. Η Κομισιόν σας ευχαριστεί που τονίζετε την ανάγκη να ενισχυθεί η διατομιακή πτυχή του προγράμματος Creative Europe κυρίως ε, για να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα των ψευδών ειδήσεων ε, μέσω του αλφαβητισμού στα μέσα ενημέρωσης. Η Κομισιόν ε, θέλει να δημιουργήσει νέα προγράμματα για να καταπολεμήσει αυτή τη μάστιγα για να κλείσω ε, κάτι για το Ευρωπαϊκό Σώμα. Το αναφέρατε κι εσείς, έγινε χθε ο τριμερής διάλογος. Η Κομισιόν επιθυμεί μια πολιτική συμφωνία το συντομότερο δυνατόν, αν είναι δυνατόν ε, τον Ιούνιο, στο δεύτερο τριμερή διάλογο, έτσι ώστε από το 18 να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο η πρόσκληση υποβολή προτάσεων για το 2018. Έτσι λοιπόν είναι κάπω επίγον το ζήτημα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εμεί θέλουμε ταχύτατη συμφωνία για το σώμα Για να εξασφαλιστεί όμω αυτή χρειάζεται και μια κάποια ευηλιξία των κρατών μελών σε σχέση με το αίτημα για νέο χρήμα. Αλλιώ δεν πρόκειται φοβούμε να υπάρξει νέα συμφωνία. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Βιώτη να πάρει και πάλι τον λόγο και μετά το Μόρτον. Παρακαλώ κύριε Βιώτη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους όσοι το λόγο. ήταν πολύ σημαντική η συζήτηση. Κράτησε σημειώσεις για τις διάφορες προτεραιότητες, ε, όπως σημειώθηκε άλλωστε συμφωνούμε σε πολλά σημεία. Δύο σκέψεις μόνο, πολύ γρήγορα. Ακόμα, είμα, περπατάμε στα τυφλά, δεν έχουμε προπολογισμό. Ακολουθούμε για τον προπολογισμό του 19 της κατευθύνης γραμμές που έχουμε ψηφίσει εκφράζουμε τις προσδοκίες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να περιμένουμε. Για το προσεχές πολιτές νομικός πλαίσιο που επίσης αναφέρθηκε. Και βεβαίω είναι αλληλεύθερα τα πράγματα, αλλά πρέπει και να τα ξεχωρίζουμε, γιατί μέχρι το 19 δεν θα έχει υλοποιηθεί το Brexit Άρα πρέπει να είμαστε σε θέση να ε, κάνουμε τις προβλέψεις μας και να δουλέψουμε πάνω σε δύο διαφορετικά επίπεδα παράλληλα και για διαφορετικές αρμοδιότητες κτλ. Για τα πιλωτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που επίσης αναφέρθηκαν, στόχος μου είναι, μια και Πρέπει να το πω, έχω τρέφω τεράστιο σεβασμό προς το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πιλωτικά έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Με ρόλος μου όμως είναι να πρόσπαστα το έργο και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με κάθε σεβασμό λοιπόν στις θέσεις και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις χρηματοδοτήσεις που έχουν χαρακτήρα τεχνοκρατικό, νομικό, κάνουν οικονομικό απαλλαγισμό, αλλά εγώ έχω καθήκον να ακολουθήσω τις οδηγίες του Κοινοβουλίου που στόχο έχει να συνεχιστούν κάποια έργα πιλωτικά που μπορεί σε όρους νομικούς, τεχνοκρατικούς, οικονομικούς να μην έχουν πάρει την υψηλότερη βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά το Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει να τα προωθήσει γιατί θεωρεί ότι υπηρετούν τους πολίτες και το δημόσιο αγαθό για τον Μακρόν και τα λόγια που εκφώνησε ίσως αφαιρέθηκα κάποια στιγμή, αλλά μάλλον εννοούσατε ότι υποσχέθηκε περισσότερη κοινωνική αλληλεγγύη ο πρόεδρος Μακρόν και περισσότερη χρηματοδότηση της κοινωνικής αλληλεγγύης με την ομιλία που εκφώνησε στο Στρασβούργο. Με χαρά άκουσα αυτά τα λόγια εγώ. Περιμένω να δω και την ε, μετάφρασή τους σε, από τα έργα. Και ελπίζω στον προσοχή προϋπολογισμό να το δούμε αυτό με Λουπίτα. Με αυτά, επιτρέψτε μου ολοκληρώνοντας να απευθύνω έκκληση και πρόσκληση προς όλες και όλους σας για συνεργασία. Ξέρουμε ότι πολύ συχνά, σχεδόν πάντα, α, όχι, ήθελα να πω εντωμεταξύ, ότι είστε τυχεροί και σαν Επιτροπή, γιατί είστε και η Επιτροπή στην οποία συμμετέχει η συνάδελφο Νίριαντ που είναι και στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών με την οποία έχουμε άμεση συνεργασία και μπορείτε όποτε θέλετε μέσω της κυρίας Νίριαντ να μου τραβάτε τα. Ε, εν πάση περιπτώσει όμω, θέλω να πω ότι ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμό μέσα στο Κοινοβούλιο δεν προξενεί αντιπαραθέσει. Σχεδόν ποτέ γιατί έχουμε κοινού στόχου. Όμω είναι σχεδόν πάντα πεδίο αντιπαραθέσεων με το Συμβούλιο. Αρχηγοί, και, κρατών και κυβερνήσεων, Υπουργοί των Οικονομικών και τη Εθνική Οικονομία, όπου έχετε εσεί κάποιο πάτημα ή κάποιο φίλο, αυτό ήθελα να πω, μιλήστε του. Έτσι, μια γλυκιά πίεση α ασκηθεί προ ε, όποιου συμμάχου μπορούμε να έχουμε στο Συμβούλιο. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διώτη. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα και που μας παρουσιάσατε αυτές τις ειδήσει. Ελπίζω να περάσει από τα λόγια στο χαρτί και να καταφέρουμε να το εφαρμόσουμε να εγκριθεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμότατα που ήρθατε σήμερα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε θα δώσω το λόγο στον Μόρτεν Λόκεργκαρ, τον εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Κύριε Διώτη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε για το χρόνο σας. Λίγα σχόλια έχω μόνο. Πρώτα, νομίζω πως ε, επισημάνθηκε πολύ σωστά ότι τα ερχόμενα χρόνια πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα έτσι ώστε οι πολίτες, ε, οι γειτονές μας να κατανοήσουν ακόμα περισσότερο τη σημασία του πολιτισμού. Είμαι μέλος της Επιτροπής για πολλά χρόνια και νομίζω πως ένα από τα κυριότερα προβλήματα που είχαμε είναι να δώσουμε στους πολίτες να καταλάβουν πόσο σημαντικός είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι το 6% του ΑΕΠ της Ευρώπης και πρόσφατα μάλιστα μιλούσαμε εκπροσώπους από το χώρο του αθλητισμού και μου είπαν ότι το 2,4% του ΑΕΠ αφορά αθλητικές δραστηριότητες. Είναι πολύ ε, μεγάλα ποσοστά αυτά, πολλά χρήματα και πρέπει να αποφύγουμε αυτές τις επιθέσεις ε, στον προϋπολογισμό μας. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιες επιθέσεις από τους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών κατά του προϋπολογισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει ο καθένας μας να συνεισφέρει όσο μπορεί. Και χάρηκα πολύ που άκουσα από την κυρία Πρόεδρο για αυτό το πρόγραμμα του Άρτε και θα το λάβουμε φυσικά υπόψη στην γνωμοδότηση. Αυτά από μένα προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Όπως και παλιότερα, έτσι και τώρα η Επιτροπή Πολιτισμού θα συνεργαστεί, θα συνεργαστεί πολύ στενά και θα αντιδράσει με μία φωνή. σε όλες τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει προς τα αγαθά τα οποία είναι τόσο σημαντικά προς όλες τις επιθέσεις του Συμβουλίου. Για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ήδη είπαμε ε, και τα πράγματα και για το Creative Europe θα χρειαστεί να πολεμήσουμε για να το κρατήσουμε, καθώς και για το εράσμος Plus. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα ικανοποιηθούμε με ένα διπλασιασμό του προπολογισμού, αλλά όπως ψηφίσαμε με μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, με τουλάχιστον τριπλασιασμό του περιπολογισμού για το μέλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμότατα και να σας υπενθυμίσω ότι η καταληκτική ημερομηνία για τροπολογίες είναι η 2η Μαΐου στις 11 το πρωί. Για την έκθεση του κυρίου Λόκεγκαρτ θα ψηφίσουμε στις 17 Ιουνίου. Μετά θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, συγκεκριμένα νούμερα και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την διαδικασία προϋπολογισμού με περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, τα δύο τελευταία σημεία της ημερήσιας διάταξης τα συνδέσαμε έτσι με πολύ κόμψο τρόπο και τώρα μας μένει μόνο το τελευταίο σημείο. Να σας ενημερώσω δηλαδή ότι η επόμενη συνάντησή μας θα είναι την Τετάρτη ε, στις 16 ε, Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 και από τις 2.30 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα και την 5η 17 Μαΐου από τις 9 μέχρι τις 12.30 το πρωί. Ελπίζω να σας ξαναδώ όλους τότε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ και τους διερμηνείς οι οποίοι έχουν εργαστεί πολύ καλά όπως πάντα.